για την αδήλωτη εργασία. Ο κύριος Πυρίνσκι έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο, ευχαριστώ και την Πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές όπως επίσης και τους φίλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία για μια επικοδομητική στάση που μας βοήθησαν να προετοιμάσουμε αυτή την πρόταση απόφασης. Η αδήλωτη αργασία έχει πολλές μορφές. Είναι κάτι το οποίο αρνείται να δώσει στους εργαζομένους τα βασικά τους δικαιώματα τους δημιουργεί συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης, δημιουργεί προβλήματα στρέβλωσης στις αγορές και γενικά ανισότητες ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στις χώρες. Είναι κάτι επίσης το οποίο αρνείται να δώσει ε, στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης όπως και στο φορολογικά συστήματα της κάθε χώρας τα απαιτούμενα. Η ανάγκη για τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας είναι κάτι το ιδιαίτερα επίγον. Λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται ε, και στην κινητικότητα των εργαζομένων και στην κινητικότητα των πολιτών γενικά. Είναι κάτι που έχει σχέση και με την ίδια τη συνέχιση της ύπαρξης της Ένωσης. Αυτή η αίσθηση του κατεπήγοντος την μοιραζόμαστε και εμείς το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως η Προεδρία. Και έτσι νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια επικοδομητική πρόταση συμφωνίας την οποία συζητάμε σήμερα. Η συμβιβαστική αυτή λύση καλεί όλες τις χώρες να είναι υπεύθυνα μέλη της πλατφόρμας είναι ένα σύστημα η πλατφόρμα αυτή που δίνει τη δυνατότητα στις χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν τα περίπλοκα προβλήματα που δημιουργεί η αδήλωτη εργασία μέσω της συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και με την συμμετοχή σαν παρατηρητών πολλών οργανώσεων και υπηρεσιών. Στόχος της πλατφόρμας καθορίζεται ε, ένα στόχος πρόληψης αποτροπής αλλά και ταυτόχρονα προώθησης μετατροπής των αδήλωτων θέσεων απασχόλησης σε επίσημες θέσεις απασχόλησης. Η αρχή της επικουρικότητας από μόνη της δεν αρκεί, αλλά παρόλα αυτά δίδεται η δυνατότητα για τη σωστή πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών, λύσεων, έτσι ώστε επιτέλους η μάστιγα αυτή να αντιμετωπιστεί. Οι δραστηριότητε της πλατφόρμα αυτής περιλαμβάνει μια, περιλαμβάνουν μια ολόκληρη σειρά συγκεκριμένων δράσεων από πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών. Έτσι τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύνολο του οπλοστασίου που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστηκαν κάποιες αμφιβολίες για το αν η πλατφόρμα αυτή είναι κάτι το απαραίτητο και για το αν δημιουργεί προβλήματα και είναι παρεμβατική στις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις επιφυλάξεις αυτές και πράγματι τις εξετάσαμε ιδιαίτερως προσεκτικά και τελικά καταλήγουμε στην πρόταση την οποία κάνουμε σήμερα. Ελπίζουμε ιδέα αποδεκτή πρόταση. Τώρα λοιπόν εμείς δεσμευόμεθα να αναλάβουμε κοινέ προσπάθειες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αδικίες που δημιουργούν οι συνθήκες της αδήλωτης απασχόλησης. Έτσι θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους, έτσι θα προστατεύσουμε τις αγορές από στρεβλό ανταγωνισμό, από τον στρεβλό ανταγωνισμό και ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε τα απαιτούμενα εισοδήματα για τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Στην ουσία στοχεύουμε στον σεβασμό του ε, κράτους δικαίου και έτσι θα αντιμετωπίσουμε το νόμο της ζούγκλας. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι. Τώρα από την πλευρά της Επιτροπής ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. οι επιτροπιστέ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, μια πιο δίκαιη ε, εσωτερική αγορά και η καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ αποτελούν για μένα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόλυτε προτεραιότητε. Προσωπικά δεν μου αρέσει ο όρο κοινωνικό ντάμπινγκ. Μιλάμε για κόσμο, δεν μιλάμε για προϊόντα, για αγαθά. Αλλά όταν μιλάμε για δήλωτη εργασία, α μην ε, καλύπτουμε με όμορφες λέξεις ε, την, ε, το μεγάλο αντίκτυπο. Η αδήλωτη εργασία λοιπόν επηρεάζει όλους τους, ε, τα επίπεδα εργασίας, την ποιότητα, τα ωράρια, την υγεία, τους όρους εργασίας, χωρίς να υπάρχει προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο κόσμος παίρνει μισθούς κρυφούς ή στο χέρι μόνο και σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρώνεται καν μετά από μήνες σκληρής δουλειάς. Μπορεί να μην έχει ε, δικαίωμα σε επιδοτήματα, σε, επιδο... σε επιδόματα ανεργίας ή απόλυση σε συνταξιωτικά δικαιώματα και το καθεξής. Η αντίρρητη εργασία δεν είναι μόνο άδικη για τα άτομα που εργάζονται σε αυτήν, αλλά και προς τις επιχειρήσεις που ακολουθούν το γράμμα του νόμου και ξέρουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι πρώτες που πλήττονται από τέτοιον άδικο και αθέμητο ανταγωνισμό και επίσης υποσκάπτει τη βιωσιμότητα του δημοσιονομικού συστήματος ε, και της κοινωνικής ασφάλισης καθότι δεν ε, δίδονται εισφορές από τις ε, αντίλετες αυτές δραστηριότητες. Είναι κρυφή η αδηλωτή εργασία και δεν μπορεί λοιπόν να προσμετρηθεί επακριβώς. Ξέρουμε όμως ότι είναι ευρεία κλίμακα σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι δύσκολο να εκριζωθεί και πως υπολογίζεται ότι αυτή η σκιώδης οικονομία φτάνει το 15 έως 20% της συνολικής οικονομίας στα, σε κάποια κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας ε, πρόληψη τη αντίληψη εργασία, Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτό το εργαλείο και τόσο σημαντικό αυτό το βήμα. Θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, ανάπτυξη ε, εμπειρογνωμοσύνη και διεξαγωγή αναλύσεων σε ό,τι αφορά επίση ε, την ε, κατάρτιση καινοτόμων στρατηγικών αντιμετώπιση και θα συμβάλλει σε μια οριζόντια κατανόηση του θέματος προβλέπεται μια πολυτομιακή προσέγγιση που θα συνενώσει διάφορες, ε, διάφορους κλάδους εμπειρογνωμοσύνης όπως είναι τα θέματα εργασιακού δικαίου, φορολογικού δικαίου και αυτή η πολυτομιακή προσέγγιση έχει ήδη εφαρμοστεί με πολύ καλά αποτελέσματα σε κάποια κράτη-μέλη και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα λοιπόν βασίστηκε σε αυτά τα καλά παραδείγματα. Μόνο μέσω μιας συνολικής προσέγγισης διασυνοριακής και διατομιακής θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πολύ αυτό φαινόμενο. Και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της συμπερίληψης ε, της πλασματικής αυτοαπασχόλησης στην πλατφόρμα αυτή, γιατί και εδώ πρόκειται για ένα τομέα όπου χρειάζεται ανάπτυξη εμπορικονομοσύνης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Τέλος. Με ικανοποίηση υπογραμμίζω ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πλατφόρμα αυτή οι κοινωνικοί εταίροι. Και η Eurofound και η OSA θα διδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλε τι προσπάθειε που έχει καταβάλει για να μπορέσει να περάσει μια ε, γρήγορη συμφωνία για την πλατφόρμα αυτή και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι και την κυρία Ουλσκοκ που προείδρευσε του τριμερούς διαλόγου τόσο αποτελεσματικά και επικοδομητικά. Σας ευχαριστώ όλους για τις προσπάθειες και για την επικοδομητική προσέγγιση το Συμβούλιο θα υιοθετήσει την απόφασή του στις 24 Φεβρουαρίου για την πλατφόρμα και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την επίσημη υπογραφή. Ελπίζω να γίνει αυτό τον Μάρτιο στην Ολομέλεια. Εν τω μεταξύ, προτιμόζομαστε για την πρώτη συνάντηση της πλατφόρμας πριν το καλοκαίρι. Και είμαι δεσμευμένη και προτίθεμαι να κάνω τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι μου, προκειμένου να σταθεί με επιτυχία η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα σας ενημερώνει τακτικά για τις δραστηριότητές της και θα υποβάλει τα προγράμματα εργασίας και τις εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και υπολογίζω στα χρήσιμα σχόλιά σας και στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Πρόεδρο. Uh, ευχαριστώ. Ε, ονόματο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, ο κ. Ντεγιόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ θετικό που έχουμε αυτή την πλατφόρμα. Μια τέτοια μορφή εκμετάλλευση όπω είναι η εργασία δεν ταιριάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανέφερε και η ε, Επίτροπο ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε και τον θέμα τον ανταγωνισμό αυτών των ε, επιχειρήσεων. Γενικά υπονομεύεται και η λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Χαίρομαι που πολλέ από τι προτάσει τη ε, επιτροπή εσωτερική αγορά έχουν ληφθεί υπόψη. Βεβαίω δεν εκπροσωπείται αυτομάτω το Κοινοβούλιο στην πλατφόρμα, γι' αυτό ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αιτήσια βάση να υποβάλει εκθέσει στο Κοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα επίση να έχει και επιχειρησιακή συνεργασία και να την προωθεί αυτή η πλατφόρμα. Όμω δεν προβλέπεται ρητός. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ορίζουν ένα εκπρόσωπο, αλλά δεν υποχρεούνται να ακολουθούν όλες ε, τις ε, διαδικασίες της ε, πλατφόρμας. Εύχομαι καλή επιτυχία λοιπόν στην λειτουργία της πλατφόρμας. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γενικών, κύριε Κούνεβα. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, η επισφαλής εργασία χειροτέρεψε πολύ στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οι ανεύθυνοι εργοδότες εκβιάζουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη να δουλέψουν και ο φόβος της ενεργίας σμπρώχνει εργαζόμενους να δουλεύουν σε συνθήκες παρανομής. Η πλατφόρμα για την καταπόλεμηση της αδειότητας εργασίας θα προσπαθήσει να βάλει μια τάξη στη τζούγκλα της της εργασίας. Καταρχά είναι σημαντική επέκταση του ρόλου της πλατφόρμας. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει ως αντίλωτη εργασία κάτι νόμιμη εργασία που δεν δηλωνόταν στις επίσημες κρατικές αρχές. Η αντίλωτη εργασία όμως παίρνει πλέον πάρα πολλές μορφές απασχόληση που δηλώνονται ως πεντάωρο, αλλά στην πραγματικότητα είναι οκτάωρο. Οι υπερορίες που γίνονται αλλά ουδέποτε πληρώνονται ψευδής αυτοαπασχόληση κλοπή των εισφορών μέχρι και το ακραίο φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας. η πλατφόρμα είναι πλέον υποχρεωμένη να τα δει όλα αυτά. τα κράτη μέλη η ευρωπαϊκή επιτροπή εργοδότες και εργαζόμενοι μαζί με τους οργανισμούς που ασχολούνται με την απασχόληση θα κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι για να κατανοήσουν την κατάσταση της εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα που επικρατεί η ισοστρέφεια και επενέρχονται ο εθνικισμός είναι κρίσιμο να ακούμε και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, το προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε κοινέ δράσεις για την καταπολέμηση της διασονοριακής αντιότητας εργασίας. Είναι αυτά αρκετά. Εμείς θέλαμε αυστηρές υποχρεωτικές δράσεις που να επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι επιπλέον που δεν συμπεριλήφθηκε μια εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων ως παρατηρητής της εργασίας της πλατφόρμας. Πιστεύουμε πως οι γυναικοί φορείς τα εισακούνται κάθε φορά που τα έχουν να συνεισφέρουν με την εμπειρία και τις προτάσεις τους. Δεν συμβαζόμαστε, απλώς τώρα ξεκινάμε. Θέλω να πω στον εισηγητή μας, τον Γιώργη Πύρινσκι, ήταν υπόδειγμα διαπραγματευτή. Θέλω να επισυνέσω και τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία και να πω πως όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στο ίδιο σκοπό και δουλεύουν με αποφασιστικότητα μπορεί να μην καταφέρουν όλα όσα ήθελαν αλλά σίγουρα δυσκολεύουν τον δρόμο των παραβατών. Καλή δύναμη σε όλους και δεν σταματάμε εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Τόμτ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα κυρία Τάισεν, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι. Η αδήλωτη εργασία είναι σίγουρα ένα από τα πιο φλέγοντα προβλήματα ε, στην Ευρώπη που ενέχει και πολλές δημοσιονομικές προπτικές. Πέραν τούτου όμως υπάρχουν προεκτάσεις ε, και για τους εργαζόμενους που πλήττονται από την αδειλωτή εργασία. Το κοινωνικό ντάμπινγκ σήμερα στην Ευρώπη είναι μια απαράδεκτη πρακτική. Όμως ε, οι κυβερνήσεις, κατά κύριο λόγο, είναι αυτές που ευθύνονται για την, και είναι υπεύθυνε για την πρόληψη και αποφυγή της αδειλωτής εργασίας στις χώρες τους. Όσοι υπό διάφορες συνθήκες ε, και υποπίεση αναγκάζονται να συμφωνήσουν, συνήθως δεν γνωρίζουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της αθλητικής εργασίας. Και έτσι αυτές οι μακροχρόνιες ε, επιπτώσεις είναι πολύ πιο σοβαρές από ότι ένα ε, βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος ε, που διευκολύνει την επιβίωση. Όμως, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν πολλές μορφές αντίλατης εργασίας και ακολουθούνται και διάφορες προσεγγίσεις για την καταπολέμησή της. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επομένως πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινή προσέγγιση και κατευθυντήρες γραμμές για την ε, πρόληψη και αποφυγή της αδίλωτης εργασίας και η πλατφόρμα είναι κατάλληλη απάντηση. Είμαι υπέρ της συμπερίληψης των κοινωνικών εταίρων, όμως είναι εξίσου σημαντικό να αξιοποιήσουμε και να τηρήσουμε την αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή, τον κύριο Περίνσκι, μετά από μακροχρόνιες ε, και δύσκολες διαπραγματεύσεις καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ κυρία και για 1,5 λεπτό. Ναι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γεώργη Πυρίνσικα και όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή και σε τελική ανάλυση είναι τεράστια η συνέπεια της αντίλωτης αυτής εργασίας στον οικονομικό κλάδο και είναι μαζικό το φαινόμενο. Αυτό έχει συνέπειες και για τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να εργαστούν με θεμητό τρόπο αλλά και για τους εργαζόμενους. Με την πλατφόρμα λοιπόν αυτή πριν από την πλατφόρμα αυτή, λοιπόν, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπήρχε ουσιαστικά σχεδόν καμία πρωτοβουλία για την ε, αντιμετώπιση τη αντίληψη εργασία, παρά το γεγονό ότι ζούμε σε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασία και κοιτώντα τι εθνικέ, του εθνικού ελέγχου εργασία, οι αρμοδιότητε του καθενό σταματάνε, σταματούσαν στα σύνορα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρώτο βήμα, σύμφωνοι, αλλά ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Και σύμφωνα με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ, ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ δεσμευτικό χαρακτήρα στην αντιμετώπιση τη αντίρρηση εργασία. Έχουμε θέματα εντοπισμού ε, επιχειρήσεων γραμματοκιβωτίων σε ό,τι αφορά τους ε, ελέγχους επίσης σε διασυνοριακό επίπεδο. Είναι καλό το γεγονός ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να δεσμεύονται να συμμετέχουν στην πλατφόρμα και είναι καλά το γεγονός ότι τα συνδικάτα τα οποία σήμερα σε πολλές περιπτώσεις καλύπτουν το πρόβλημα της ε, ε, εργασίας συμμετέχουν. Αλλά χρειαζόμαστε πανευρωπαϊκούς ε, κανόνες και διασυνοριακή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μακιντάιρ για δύο λεπτά. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι, να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις για μια εξαιρετική δουλειά. Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι αυτό ωφέλισε το Κοινοβούλιο. Η αδήλωτη απασχόληση είναι σοβαρότατο θέμα. Επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη, επηρεάζει τα φορολογικά έσοδα, δημιουργούνται προβλήματα από τη φοροαποφυγή, απάτες στο σύστημα προστασίας της εργασίας, την παράνομη μετανάστευση και φυσικά υπονομεύει και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η πλατφόρμα αυτή λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το ευρωπαϊκό ε, δεδομένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέμβει. Δίδει προστιθέμενη αξία μέσω της δυνατότητας ανταλλαγής επιρριών βέλτιστων πρακτικών και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην βελτίωση μέσω αυτής της πλατφόρμας ενώ της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών αναγνωρίζοντας πάντα βέβαια την εθνική τους κυριαρχία. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι το επίπεδο της αδήλωτης εργασίας ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με κάποια δεδομένα του ΩΣΑ, η ανεπίσημη εργασία είναι 1,7% ενώ σε άλλες χώρες αυτό γίνεται 30%. Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες. Καταρχάς, η εμβέλεια της πλατφόρμας θα περιοριστεί στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Και όχι, η πλατφόρμα δεν έχει σαν στόχο να επιβάλλει ενιαίες απόψεις πρέπει να υπάρξει σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Η συμμετοχή βέβαια στην πλατφόρμα είναι υποχρεωτική, αλλά οι δραστηριότητες ε, θα είναι σε θελοντική κατά περίπτωση βάση. Είναι ένα καλό μέτρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μακιντάρη, έχετε δύο μπλε κάρτες, Χιρσάνη και Εύριτς. Τις αποδέχεστε? Ναι, ωραία. Κύριο Σάνι πρώτα. Παρακαλώ τηρήστε το χρονικό όριο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Κύριε Μάκιντάιρ, αν σωστά κατάλαβα αυτά που είπατε, η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί σε θέματα συνεργασίας και να μην έχει ε, δεσμευτικούς ε, κανόνες, αλλά πολλοί θεωρούν αυτονόητο ότι η εισαγωγή ενός ενιαίου κατώτατου μισθού στην Ευρώπη θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη. Το υποστηρίζετε λοιπόν αυτό. Εσείς ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μακιντάρη για να απαντήσει. Α, συγγνώμη, να ακούσουμε και τη δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ και καλημέρα και στους συναδέλφους. Είπατε ότι θα πρέπει κάποιες χώρες να συνεργαστούν σε ό,τι αφορά τα θέματα της εφαρμογής. Νομίζω το είπε και ένας άλλος συνάδελφος αυτός. Υπάρχει οποιοδήποτε λόγος γιατί κάποια από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρατε, τα οποία είναι λογικά και σωστά, θα μπορούσαν να γίνουν από ένα ανεξάρτητο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια ελεύθερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά σε μια συμφωνία απλή συνεργασία. Η κυρία Μάκιντάρ για να απαντήσει τώρα. Ευχαριστώ. Απαντώντας την πρώτη ερώτηση. Ο ελάχιστος μισθός δεν έχει καμία σχέση με την πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία. Ίσως παρανοήσατε τα λεγόμενά μου. Ε, ε, υπάρχουν διαφορετικές ενέργειες τις οποίες μπορεί να κάνει η πλατφόρμα και κάθε μία από αυτές θα είναι εθελοντική. Τα κράτη-μέλη θα επιλέγουν ποιες πλευρές έχουν σημασία για αυτές. Η ενισχυμένη συνεργασία είναι ένας καλός τρόπος, θα έλεγα, από κοινού αντιμετώπισης του προβλήματος. Τώρα για τη μόχλευση. Προφανώς τώρα από το δικό σας κόμμα εσείς δεν θέλετε να υπάρχει τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ διαφέρω. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις και αυτή είναι μία από αυτές όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει αξία στην προσπάθειά μας και γι' αυτός θα ήθελα να συμμετέχουμε τόσο το καλύτερο που όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν εδώ έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την αδήλωτη εργασία η οποία είναι άλλωστε διασυνοριακό φαινόμενο. Αν θέλετε τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο να δημιουργήσετε τη δική σας οργάνωση θα έχετε περισσότερες δυσκολίες γιατί δεν θα έχετε τους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας με τις υπόλοιπες χώρες με ισότιμο τρόπο. Thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Πυρίνσκι και τους κοιόδης εισηγητές και το Γιάννη Τσούμ από τη δική μας πλευρά για την πλήρη εφοσίωσή τους και δέσμευσή τους να διασφαλίσουν ότι θα καταφέρουμε να συστήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα ενισχύσει τη συνεργασία στην πρόληψη και αποτροπή της αδειλωτής εργασίας. Το γεγονός ότι η συμμετοχή είναι υποχρεωτική σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη υποχρεωτικά πρέπει να συμμετάσχουν. Και επομένω θα πρέπει να εμπλεκούν και στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνη και αναλύσεων. Και αυτό από μόνο του θα συμβάλλει σε μια οριζόντια κατανόηση όλων των ζητημάτων που συνδέονται με την εργασία. Ωστόσο, ενώ η συμμετοχή είναι υποχρεωτική, οποιασδήποτε συστάσεις για ανάληψη δράσης που στηρίζονται από την ε, πλατφόρμα ε, εφαρμόζονται σε θελοντική βάση από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έχοντας συμμετάσχει στην ανάπτυξη εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση αδήλωτης εργασίας. Αυτά τα κράτη-μέλη λοιπόν που τα έχουν κάνει όλα αυτά έχουν πολύ πιο πιθανότητες να εφαρμόσουν κιόλα αυτές τις ε, πρακτικές ε, της ε, πλατφόρμας. Δεν θα προτείνει πλατφόρμα εναρμόνιση των νόμων, αλλά θα παράσχει πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Στα 18% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ αν έρχεται εργασία και πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι αρνητικέ οι επιπτώσει και για του εργαζομένου, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό τη. Πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε ευάλωτη εργασία, πολύ συχνά αποδέχονται πολύ κακέ εργασίες, εργασία, χωρί χωρίς καμία ε, ασφαλιστική σφορά, ασφάλιση, ε, περιθάλψη, επισφαλή εργασία ενώ η κοινωνία χάνει έσοδα από φόρου, από ασφαλιστικέ φορέ και υπάρχει και ο θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Στην επόμενη συζήτηση θα εξετάσουμε το φορολογικό πακέτο για την φοροαποφυγή που απαιτεί συντονισμένη δράση. Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρχει τέτοια συντονισμένη συνεργασία υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα λειτουργήσει σε εθνικό και σε διασυνορικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Κάρη, για ένα λεπτό. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια για την προσπάθεια την οποία έκαναν. Είδαμε στο εσωτερικό της ενίας αγοράς να υπάρχουν πολλές κοινωνικές αλλαγές. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ένα τρομερό ανταγωνισμό σε εργασιακό επίπεδο. Αυτό οδηγεί ουσιαστικά προς την αδήλωτη εργασία. Αυτό φυσικά είναι αρνητικό για τον εργαζόμενο, αλλά και για την κοινωνία που χάνει αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης και χάνει και φορολογικά έσοδα. Συνεπώς η πρωτοβουλία αυτή είναι μια θετική πρωτοβουλία για περισσότερες μορφές συνεργασίας και συντονισμού. Αλλά νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα και οφείλουν να ασκήσουν αυστηρότερους ελέγχους όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αναφέρομαι στην Νορβηγία σαν παράδειγμα, όπου μπορεί να υπάρχουν έλεγχοι από τους επιθεωρητές εργασίας αλλά γίνονται και προσπάθειες ευαισθητοποίησης των ίδιων των εργαζομένων. Η κυρία Νούκια για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Πυρίνσκι, αγαπητοί σκιώδες συζητητέ. Η αδέλωτη εργασία είναι πολύ μεγάλο αλλά συχνά αόρατο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελέτε δείχνουν ότι ο άτυπο ε, τομέα φτάνει το 18,4% του ΑΕΠ στα κράτη μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει πολλέ αρνητικέ προεκτάσει. Δημιουργεί ε, τεράστιε φορολογικέ απώλειε, αθέμητο ανταγωνισμό και τιμωρεί ουσιαστικά τους εργοδότε ε, που τηρούν το γράμμα του νόμου και απασχολούν τους εργαζομένους υπό δίκαιες συνθήκες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι εκμεταλλεύεται τους εργαζομένους ε, και υπονομεύει τα δικαιώματά τους και την κοινωνική τους ασφάλιση. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την αδηλωτή εργασία και αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μα, πρέπει να το καταπολεμήσουμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε αυτή την πλατφόρμα κάνουμε το πρώτο βήμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ε, για την ενημέρωση των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να πάρουν πιο αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Γιατί αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το θεμητό ανταγωνισμό, την κοινωνική ασφάλιση και τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ως αφετερία μόνο αυτή την πλατφόρμα για να διαμορφώσουμε πιο συντονισμένες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είτε είναι ε, ο συντονισμός εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ε, ε, η επιβολή κυρώσεων στου εργοδότε που εκμεταλλεύονται αυτό το φαινόμενο τη αδέλφου εργασία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί η αδέλφου εργασία είναι μία από αυτέ τι μεγάλε ευρωπαϊκέ προκλήσει. Α αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή την πλατφόρμα για να αντιμετωπίσουμε την αδέλφου εργασία και για να κάνουμε βήματα για να διαμορφώσουμε ένα υγιέ ε, από κοινωνική άποψη οικοδόμημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κόλλινς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Οι μοναδικές θέσεις απασχόλησης που βλέπουμε ότι δημιουργούνται είναι ε, τέτοιες ε, θέσεις απασχόλησης όπως ε, σε τέτοιες πλατφόρμες όπου δημόσιοι υπάλληλοι, εθνικές, εθνικοί φορείς και άλλοι αντίστοιχοι φορείς που λαμβάνουν και συνδρομή από κάποιες γραμματείες, έτσι μαζεύονται και τα λένε. Ακούμε πολλά για επιχειρήσει που φοροδιαφεύγουν. Πολλέ από αυτές βέβαια προέρχονται από την περιοχή του Λουξεμβούργου, όπου ο ίδιος μας ο πρόεδρος, ο Γιούγκερ, ήταν πρωθυπουργό για 15 χρόνια. Όμω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η φοροαποφυγή, σε αντίθεση με την φοροδιαφυγή, δεν είναι παράνομη, παρότι πολλοί, ιδίω όσοι δεν έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, ε, και να έχουν παράλληλα μαύρα ταμεία ε, δυσκολεύονται ε, να ξέρουν να μάθουν διαφορά. Οι ιδιωτικέ επιχειρήσει αξιοποιούν καλύτερα όμω τα χρήματά του από ό,τι θα κάνει ποτέ μια δημόσια επιχείρηση. Αν είχαμε όμως οικονομικές προβλέψεις ε, που ε, να στηρίζουν τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ο George Osborne, δεν θα υπήρχε ανάγκη για, ούτε για φοροαποφυγή, ούτε για δήλωτη εργασία, ούτε για επανόμευση της κοινωνικής ασφάλισης. Όμως αυτό είναι ε, διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων. Όμως έχουμε βρει χρήματα παρά το τεράστιο χρέος για να δώσουμε 250 εκατομμύρια κάθε χρόνο ε, σε αυτή την πλατφόρμα να κατασπαταληθεί σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια και σε αεροπορικά εισιτήρια. Βλέπουμε ότι η απορρίθμιση είναι αυτή ε, που προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει λοιπόν να καταργήσουμε αυτό το, ε, το γελίο όμιλο συζητήσεων και αφού ξεκινάμε α κάνουμε το ίδιο και στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στο Λουξεμβούργο και θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Thank you. Uh, Mr. two minutes. Ευχαριστώ κύριε Μαχτάν για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Βεβαίω πρέπει να αποθαρρύνουμε και να αποτρέψουμε την αδειλώτη εργασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο χάρη σε μια πλατφόρμα που θα συγκεράσει τα, όλα τα κράτη-μέλη. Όμω ε, πρέπει να εξετάσουμε και άλλα ζητήματα. Πρώτον θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιε είναι οι αιτίε τη αδειλώτη εργασία. Έχουμε έναν εργοδότη και έναν εργαζόμενο από την άλλη και οι δύο συμφωνούν για να μην πληρώσουν καμία εισφορά, κανένα φόρο. Και αυτό γιατί, γιατί η εργασία δεν επιτρέπει στον εργοδότη ε, να ευμερίσει και στον εργαζόμενο να επιβιώσει για να προσαρμοστούμε, όπω λέμε, στην παγκοσμιοποίηση εξαιτία των ε, φορολογικών σα ε, πολιτικών και των πολιτικών λιτότητα που ε, καταργούν χιλιάδε θέσει εργασία. Ποιε είναι οι επιλογέ ενό εργοδότη και ενό εργαζομένου. Ο εργοδότη μπορεί είτε να χαθεί, είτε να καταργήσει θέσει εργασία στη χώρα του είτε να επικαλεστεί διάφορε προκλήσει και διαδικασίε, είτε, όπω αναφέρεται στην έκθεσή σα, να μην δηλώνει την εργασία των υπαλλήλων του. Από την άλλη, ο εργοδότη με ή χωρί δουλειά μπορεί ούτε να μεταναστεύσει σε καλύτερε περιοχέ, αλλά δεν είναι απλό, είτε ε, να μπει στην ανεργία, αλλά δεν φτάνουν τα επιδόματα είτε να πάει στις διάφορες θεσισίτια για να πάρει φαγητό, να πάρει ρούχα, αλλά εντάξει για τους οικογενειάρχες αυτό είναι πολύ δύσκολο, είτε να εργαστεί στα μαύρα, μόνο και μόνο για να γεμίσει το ψυγείο του. Κατανοούμε λοιπόν ότι η πλατφόρμα σας δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Και με την τεράστια ε, μαζική εισρωή των ε, προσφύγων που θέλετε να αποδεχθείτε και με τα όσα προβλέπονται και στον ΠΟΕ. Πρέπει να διαμορφωθεί μία πολιτική οικονομικής ανάπτυξης ε, με έναν έξυπνο ε, προστατευτισμό και βοήθεια προς τις επενδύσεις. Ε, Ο κύριος Ζαγιανόπουλος για 1,5 λεπτό. Όταν η αδίλωτη εργασία σε όλη την Ένωση οργιάζει στο 20%, ενώ στην ελλάδα ξεπερνά το 36% και σε κερδοφόρους κλάδους όπως ο τουρισμός το 44% χτυπώντας ιδιαίτερα γυναίκες και νέους και η βασική επιδίωξη της ένωσης όπως δηλώνει είναι η μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους με απαλλαγή εργοδοσίας και κράτους από το κόστος της ασφάλισης είναι κυριολεκτικά σκέτη κοροϊδή η ανησυχία της για τη μείωση της αδείλωτης εργασίας καθώς ούτε μέτρα ασπιρίνες δεν προτείνει η πλατφόρμα την αντιμετωπίζει μόνο σαν αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων σαν όχημα για τη συμπίεση των μισθών σαν κίνητρο για μερική μετατροπή της μαύρης εργασίας σε ευέλικτη εργασία μερική και εκπεριτροπής απασχόληση μπλοκάκια εκμετάλλευση της μαθητείας κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα δουλεμπορικά γραφεία. βέβαια η μαύρη εργασία θα συνεχίσει να υπάρχει γιατί συμφέρει στο σύστημά σα. για παράδειγμα στην ελλάδα η αύξηση ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών στο 75% του συνολικού εισοδήματο σε αυτοαπασχολούμενου και αγρότε, με το νέο σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θα αυξήσει την αδήλωτη εργασία, θα του απομακρύνει από την ασφάλιση, τη σύνταξη και την περίθαλψη. Η νέα γενική μείωση μισθών και εργοδοτικών εισφορών, η αύξηση τη ανεργία είναι τα φόπλακα για το ασφαλιστικό σύστημα και τα ταμεία. Απάντηση σε αυτό τον αρμαγεδόν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δίνουν ενιαία εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι φτωχοί αγρότες με την γενική τους πανελλαδική απεργία στις 4 του Φλεβάρι. Ευχαριστώ κύριε Σμάν για ένα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η μαύρη αντίλεπτη εργασία δεν ε, είναι μικρό φαινόμενο. Στη Γερμανία ε, μου και μόνο ε, πέρσι 340 δισεκατομμύρια μας κόστισε. Και όποιος λοιπόν ε, στερεί και βλάπτει έτσι την κοινωνία θα πρέπει να υπολογίσει σε ε, ποινές. Αυτό είναι σωστό. Υποστηρίζω λοιπόν την πλατφόρμα που είναι ένα υπόδειγμα για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Αντί να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε ξεχωριστά το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ευρύτερη εργασία, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν αποδεδειγμένα καλές πρακτικές από άλλες χώρες. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν από κοινού το συντονισμό των λειτουργικών μέτρων και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται από την πλατφόρμα με ένα πιο σωστό κόστος. 2,1 δισεκατομμύρια αναέτος από το Progress. Είναι σημαντικό οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής και τα εγχειρίδια να μην είναι δεσμευτικής φύσης, γιατί τα εθνικά συστήματα επιθεώρησης έτσι δεν θα επηρεαστούν. Η προηγούμενη Επιτροπή, για παράδειγμα, είχε πρόβλημα με τις επιθεωρήσεις εργασίας στη Γερμανία και μάλιστα μας είχε προσαγάγει στο δικαστήριο και έχασε. Με τον Ζαν Κλοντ Ιούγκερ και με την ε, κυρία Τάισεν θα ήθελα να πω το εξής, ότι η πράξη έχει αποδείξει ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο με υψηλό επίπεδο ελέγχου και μόνο έτσι θα υπάρχει και μια ευρεία αποδοχή και θεωρώ ότι μια καλή βάση είναι ο συμβιβασμό ο οποίος βρέθηκε πλέον στο τρομερή διάλογο και αποτελεί μια σημαντική και καλή αρχή. Ευχαριστώ η κυρία Ουλσκφοκ για ένα λεπτό, μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καταρχάς σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί η αδίλωτη εργασία οδηγεί σε σημαντικές ζημίες στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις, τα κοινωνικά επιδόματα, σε ό,τι αφορά τη φορολογία και φυσικά προκαλεί και αθέμητο ανταγωνισμό. Όσοι δεν δηλώνουν την εργασία έχουν ένα πλανέκτημα που δεν έχουν οι άλλοι. Και επίσης ε, η ιατρική εργασία συνδέεται με επισφαλείς όρους εργασίας και με τον κίνδυνο εκμετάλλευσης. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ουσιαστικά για ε, μια μορφή δουλείας. Ε, αν οι επιχειρήσεις πληρώνουν τις κοινωνικές εισφορές για τους εργαζόμενους, μάλλον χωρί τις κοινωνικές εισφορές από πλευρά των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν συνταξιδοτικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω αυτή την πλατφόρμα ως ένα πρώτο βήμα για την καταπολέμηση της εργασία και χαιρόμαστε που εκπροσωπήθηκαν στην πλατφόρμα αυτή και οι κοινωνικοί ατέροι, γιατί αυτοί συναποτελούν την αγορά εργασίας. Και νομίζω ότι έτσι θα καταστεί η πλατφόρμα ε, πολύ ε, αποτελεσματική. Αλλά ας μην εφησυχαστούμε, γιατί παράλληλα ο κόσμος μαστίζεται από τη φτώχεια. Και αυτό είναι το θέμα, προκειμένου να μην αποδέχεται οποιαδήποτε δουλειά άσχετα με το κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε διασνοριακούς κανόνες προκειμένου να μην επιτρέπεται η εκμετάλλευση του κόσμου. Να υπάρχει ίδιοι όροι και ίσοι όροι με την ίση αμοιβή και όσοι είναι θύματα εγκληματικών ενεργειών να μπορούν να απευθύνονται στο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Από τον κύριο Κάβορ έχετε μπλε κάρτα, κυρία Ουλσκούτ. Την αποδέχεστε. Αποδέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Κάβορ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που αποδέχεστε την μπλε κάρτα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα και κανεί δεν υποστηρίζει ασφαλώ την αντιλήτη εργασία, αλλά μήπω θα πρέπει να κοιτάξουμε την κατάσταση τη κοινωνία. Η φύση τη κοινωνία επιτάσσει ότι πάντα θα υπάρχει κόσμος κάτω από το κατόφλι της στόχιας και αυτός ο κόσμος θα κάνει αντιλήτη εργασία απορρίθμιση, απορρίθμιση το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό χρειάζεται. Και στην βρετανική οικονομία να δοθεί η ευκαιρία να προχωρήσει μπροστά. Γιατί η υπερβολική ρύθμιση αυτή είναι που αξιοθετεί τον κόσμο στην αδηλετή εργασία. Η απάντηση. Είναι... είναι δύσκολο να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά που αναφέρετε. Αλλά να σας πω, ότι οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, ανταγωνίζονται άλλες μικρές επιχειρήσεις με αθέμητους όρους, με αδύλατους εργαζόμενους, δεν ε, μπορούμε να μιλάμε στην περίπτωση αυτή για δίκαιους κανόνες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να. πρέπει να φροντίσουμε στο κράτος δικαίου να τιμωρούνται όσοι ακολουθούν αθέμητε πρακτικέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, κύριο Χοκ. Ευχαριστώ. Αναμφίβολα πρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της αθλητής εργασίας. Όμως, καλύτερα θα ήταν να διαμορφώναμε ένα σύστημα μέσω στο οποίο οι επιχειρήσεις να μην επιθυμούν καν να ακολουθήσουν τέτοιες πρακτικές. Επομένως, αυτή η πλατφόρμα θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για την κατάρτιση μιας στρατηγικής και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για φοροαπαλλαγές, φοροδιευκολύνσεις, ε, διευκόλυνση ε, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και κίνητρα για την απασχόληση. Με παράλληλη τήρηση και σεβασμό του εργασιακού δικαίου. Ευχαριστώ. Καλβέτ Τσαμπών, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Εγώ πιστεύω ότι η σημερινή μέρα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους εργαζομένους. Επιτέλους αναγνωρίζουμε ότι είναι ευρωπαϊκό ένα πρόβλημα το οποίο μας επηρεάζει όλους και το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σταδιακά μόνο μέσα από μια ευρωπαϊκή προοπτική. Προφανώς η μάστιγα της υπόγειας οικονομίας είναι τρομερή, δημιουργεί προβλήματα στη χρηματοδότηση της κοινωνικής απασχόλησης, στα φορολογικά έσοδα, μειώνει και υπονομεύει την ίδια την δημοκρατία γιατί καταδικάζει ανθρώπους να ζουν εκτός νόμου. Είναι κάτι το αφόρητο, κάτι το απαράδεκτο, είναι η άκρα εκμετάλλευση ε, των πιο απελπισμένων τμήματων της κοινωνίας μας. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και νομίζω ότι σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Πιμιέντα Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι πολιτικές της δεξιάς οι οποίες ακολουθούνται στην Πορτογαλία παράλληλα με αυτές τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν στην πλήρη απορρίθμιση της εργασίας και στην αμφισβήτηση των συλλογικών συμβάσεων. Συνεπώς στην Πορτογαλία καταλάβαμε πια ότι οι πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται από την Τρόικα έχουν συνεισφέρει στο να αναπτυχθούν, στο να αναυξηθούν, αυξηθούν οι περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας. Η προσφυγή επίσης σε συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης οδηγεί στην, στο να κάνει προσωρινή την απασχόληση των εργαζομένων. Η καταπολέμηση αυτής της προσωρινότητας, η καταπολέμηση της φτώχειας, η καταπολέμηση της παράνομης εργασίας δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο μέσω του σεβασμού ε, της ε, συλλογικής σύμβασης ε, κάτι το οποίο είναι αντίθετο από αυτά τα οποία επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Σόλτες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η αδήλωτη εργασία, όπως έχουν πει και πολλοί συνάδελφοι, έχουν, έχει πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς ε, τομείς, κυρίως ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα συνταξιδοτικά τους δικαιώματα, αλλά και τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Και βεβαίως έχει σημαντικές διχρονομικές ε, προεκτάσεις για τον κρατικό προπολογισμό και για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η αλήθεια είναι ότι με αυτή την πλατφόρμα, που βέβαια σίγουρα τη στηρίζουμε, πολλά ακόμα μένουν να γίνουν. Μία πτυχή είναι η φορολογική πολιτική που ουσιαστικά δεν θα υποχρεώσει τις επιχειρήσεις ε, να μην ακολουθήσουν αυτή την πρακτική. Επίσης, όσοι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς θα πρέπει να αποδείξουν ότι ακολουθούν τις απαραίτητες ε, δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των δικαιωμάτων και χρειαζόμαστε και πραγματικά στοιχεία για να ξέρουμε συγκεκριμένα τα στοιχεία σε ό,τι φορά την εργασία. Έχετε μια μπλε κάρτα, την αποδέχεστε. Όχι. Από τον κύριο Γιακοφτσίτς. Για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτες που δεχθήκατε την μπλε κάρτα. Το ερώτημά μου είναι, συμφωνείτε ότι η διαφορά μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά την παραοικονομία Βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες ε, η αδεύτερη εργασία είναι 1,2% και σε άλλες χώρες είναι 30%. Αυτό μπορεί λοιπόν μπορεί να επιληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως ε, μέσω μιας ε, ευρωπαϊκής επιθεώρησης εργασίας θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Σίγουρα. Να πιστεύω ότι η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν υπάρχει ένα ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομίζω ότι και ένα σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι και το δικαίωμα στην απασχόληση και στην αξιοπρεπή ζωή. Καλό θα ήταν λοιπόν ε, να προαγάγουμε περαιτέρω αυτή την ε, επιθεώρηση, την πλατφόρμα, με μια ευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασία, για παράδειγμα, όπω θα πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κάποιο λοιπόν, ο οποίο θα διασφαλίζει ότι η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων είναι υψηλή ποιότητα και δεν θα υπάρχει αυτή η διαφορά ε, και θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ των χωρών σε ό,τι φορά την αδελφή εργασία. Ευχαριστώ κυρία Βεγγίν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι φτάνουμε στην ψηφοφορία για την πλατφόρμα αυτή. Η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας ήταν κάτι το θετικό. Προώθησε τη συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες επιθεωρήσεις εργασίας. Αυτό θα έχει κόστος βέβαια. Θα πρέπει λοιπόν να μην πέσουμε για μια ακόμη φορά σε παγίδα και η υπηρεσία αυτή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει, δηλαδή τη μαύρη εργασία. Αυτές είναι ακραίες μορφές εκμετάλλευσης των εργαζομένων που δεν ε, ε, χτυπά μόνο τους μετανάστες αλλά και τους Ιταλούς γεωργούς και αυτό φάνηκε από τα παραδείγματα τα φρικτά που είχαμε φέτος το καλοκαίρι στην Ιταλία. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε έτσι ώστε η καταπολέμηση της μαύρης εργασίας να καταστεί ευρωπαϊκό θέμα. Κυρία Μελά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην κοινωνία μας, στη δυτική κοινωνία, οι ανθρώπινες δραστηριότητες ε, είναι πια τμήμα του εμπορίου. Αντίθετα με τις ε, βιοτεχνικές ε, δραστηριότητες η παγκοσμιοποίηση των ανταλλαγών λειτουργεί με τα κριτήρια της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας εις βάρος του σεβασμού των προσώπων. Η παγκοσμιοποίηση ε, πλέον υπερισχύει του σεβασμού των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και αμφισβητείται η ε, κυριαρχία μιας ε, χώρας να διατηρήσει υψηλής ποιοτικής τάχνης παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και δύο αιώνες από τον χριστιανικό ουμανισμό εδώ και δύο αιώνες προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και σήμερα. Δυστυχώς όμως η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί τεράστια κρυφά υπόγεια κέρδη. Το κόστος το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται ε, να παίρνουν μισθούς οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι επίγον να αντιμετωπιστεί η μαύρη εργασία γιατί η νέα ψηφιακή επανάσταση στην ουσία θα δημιουργήσει σε μια τεράστια φούσκα και απάτη. Η Ευρώπη είναι θα έλεγα σε κακή θέση για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν σε εθνικό επίπεδο να είναι αποτελεσματικά. Ναι σε μια διεθνή συνεργασία όχι σε μια υπερβολική παρέμβαση της Ευρώπης, της ανεπαρκέστατης Ευρώπης, ιδιαίτερα λόγω ε, του χαρακτήρα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην ξεχνάμε και τα 10.000 παιδιά των μεταναστών που χάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Κύριος Φουντούλης. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να σταματήσουμε τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων αποτελεί ντροπή για την ευρώπη του δύο το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας να έχει τέτοια έκταση. κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει εξασφαλισμένη κοινωνική πρόνοια ασφάλιση ένα δίκαιο μισθό και μια σύνταξη που θα του εξασφαλίζει άνετη ζωή μετά. όμως η ένωση μόνο στα λόγια ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους υποβαθμίζεται ακόμα και τα πιο βασικά δικαιώματα των εργαζομένων επικαλούμενη μια δίθεν ανταγωνιστικότητα μετατρέπετε ολόκληρες χώρες όπως η πατρίδα μου σε ειδικές οικονομικές ζώνες και έχετε το θράσος να μιλάτε για εργαζόμενους και προστασία. να έρθετε στην ελλάδα να τα πείτε αυτά στην ελλάδα όπου με τις πολιτικές σας έχετε δημιουργήσει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και ισχυρίζεστε πως αυτό είναι ο δρόμος προς το μέλλον. σας το χαρίζουμε αυτό το μέλλον εμείς αγωνιζόμαστε για το δικό μας μέλλον σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή ένωση. λέμε όχι σε μια ένωση προστάτη του μεγάλου διεθνού κεφαλαίου μια ένωση αρχιλιστή που με τις φορολογικές επιδρομές που διατάσσει και εκτελούν οι εγχώροι υποτακτικοί της επιδιώκει να καταστρέψει κάθε ίχνος εθνικής οικονομίας ώστε να μοιράσει τα συντρίμμια στις πολυεθνικές της επιπλέον όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε για τα δικαιώματα των εργαζομένων επιδιώκετε σταθερά εδώ και πολύ καιρό την αντικατάσταση της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης από τις ορδές των λαθρομεταναστών γνωρίζοντας βέβαια πόσο πιο εύκολο θα είναι να εκμεταλλευτείτε το καινούργιο αυτό εργατικό δυναμικό και να επιτύχετε μια εξομοίωση προς τα κάτω και πάλι προς το συμφέρον των πολυεθνικών άλλωστε θυμηθείτε πω ο ίδιο ο πρόεδρος σούλτς είχε ζητήσει για την ευρώπη 50 εκατομμύρια νέου μετανάστες. να ξέρετε όμως πως οι λαοί ξυπνάνε και θα στείλουν εσά και τις πολιτικές σας στα σκουπίδια της ιστορίας όπου και ανήκετε. Uh, Κύριε Φουντούλη, έχετε μπλε κάρτα από την κυρία Γκραπίνη. Τι δέχεστε? Μάλιστα, κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, είπατε μεταξύ άλλων ότι δεν θέλετε την προστασία των μεγάλων επιχειρήσεων, του μεγάλου κεφαλαίου. Συμφωνείτε όμως ότι μόνο με τη συνεργασία μεταξύ των κριτών μελών, με τη συνεργασία μπορούμε να εντοπίσουμε την αδίλωτη εργασία και να μην προστατεύουμε παραβιάσεις των εργασιακού δικαίου. Αγαπητοί συνάδελφε, μάλλον δεν καταλάβετε καλά, ήταν λάθος η μετάφραση. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα εγώ είπα ότι πρέπει να προστατεύουμε όλους τους εργαζόμενους γιατί όλοι έχουν ίσα δικαιώματα είτε δουλεύουν σε μικρές επιχειρήσεις είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις αλλά δυστυχώς με τις πολιτικές αυτές προστατεύονται οι πολυεθνικές και όχι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Thank you. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Για λεπτό σε μια μελέτη του Ευρωβαρομέτρου το 2013 η αδήλωτη απασχόληση αντιπροσώπηβε το 15 με 20% κάποιων κρατών μελών. Όλοι συνειδητοποιούμε ότι η αδήλωτη εργασία είναι μια απειλή τεράστια για τα οικονομικά μας πρότυπα. Πίσω από τον όρο παράνομη εργασία κρύβεται φυσικά η προσωρινότητα στην απασχόληση, η έλλειψη αξιοπρέπειας του εργαζομένου και η πτώση των εσόδων για την κοινωνική ασφάλιση. Η αύξηση της αδήλωτης εργασίας δημιουργεί μια αίσθηση αδικίας στους συμπολίτες μας που σέβονται τους κανόνες. Παρατηρήσαμε επίσης ότι οδηγεί ορισμένες περιοχές και κράτη στην πλήρη αποτυχία. Συνεπώς λοιπόν η πρόταση αυτή που δεν είναι μία επιπλέον νομοθετική ρύθμιση αλλά μία βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει την άκρα δεξιά στο να την υπερψηφίσει κανονικά. Δεν θα καταλάβαινα μία αρνητική στάση. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μία συντονισμένη απάντηση μην ξεχνάμε ότι η καταπολέμηση της μαύρης εργασίας θα πρέπει να γίνεται και σε επίπεδο πρόληψης. Πρέπει να το πούμε ότι πολλές φορές οι εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα των εργασιακών είναι ανεπαρκείς. Όπως δείχνει η μελέτη του Ευρωπαρομέτρου θεωρούν ότι το 50% μάλλον θεωρεί ότι ε, είναι κάτι το αρνητικό και για την οικονομία και για τους εργαζομένους. Πρέπει να καταπολεμήσουμε λοιπόν την αδήλωτη εργασία, πρέπει όμως να έχουμε σωστούς κανόνες λειτουργίας, σωστές νομικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να προχωρούν να αναπτύσσονται. Ευχαριστώ κυρία Γιονγκέριους για ένα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τους σημερινούς καιρούς Τη επιλογή μεταξύ της ανεργία, τη μαύρη εργασία ή της ε, επισφαλούς εργασία, βλέπουμε ότι ε, οι εργαζόμενοι βρίσκονται μεταξύ σκύλου, και Επομένω, Επομένως, ε, είναι θετικό που αυτά τα φαινόμενα έρχονται στο φω, και μπορούν οι εργαζόμενοι να απολάβουν τον δικαιωμάτων του, των εργασιακών του δικαιωμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την ομάδα του για την πολύ καλή αυτή προσπάθεια για τη σύσταση αυτή τη πλατφόρμα για την αντιμετώπιση τη μαύρη εργασία. Είναι ένα πρώτο βήμα στην σωστή κατεύθυνση για την ε, αντιμετώπιση τη εκμετάλλευση των εργαζομένων, τη εκμετάλλευση ε, τη κοινωνική ασφάλιση και του αθέμητου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτή η πλατφόρμα, ελπίζουμε, ε, να ενισχύσει τη συνεργασία και μεταξύ κρατών μελών Όλα αυτά είναι πολύ θετικά στοιχεία. Κάτι άλλο θετικό είναι ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ω ισότιμο μέλο τη πλατφόρμα, θα συμβάλλει στην, ε, στον προσδιορισμό των προβλημάτων σε συγκεκριμένου κλάδου, σε συγκεκριμένε χώρε. Και γι' αυτό είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν σε αυτή την προσέγγιση. Για παράδειγμα στο Βέλγιο. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε στο ότι ε, ο αρμόδιος υπουργός ε, έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τεράστια έσοδα για τα κοινωνικά ταμεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και την Επίτροπο τι συμβαίνει με την αγορά εργασίας. Γιατί μαζί με την πλατφόρμα χρειαζόμαστε και αντίστοιχη νομοθεσία για να κλείσουμε τα νομικά κενά. Thank Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Η έκθεση για την ε, ίδρυση μια ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας, για την πρόληψη της της εργασίας, της μαύρη εργασίας, αποτελεί απόρρια δύσκολων διαπραγματεύσεων και μεγάλη επιτυχία από πλευράς και προσπαθειών του ECR. Πέρασε λοιπόν επιτέλους το ότι η αποδοτικότητα των κρατών μελών στην αντιμετώπιση του φαινομένου είναι διαφορετική και αυτό θα πρέπει να επιληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό επαρκώς και θα ήταν σαφώς ανόητο να τις επιβαρύνουμε με επιπλέον κανόνες για τα κράτη-μέλη. Υποχρεούνται να συμμετέχουν και να διαβουλεύονται στην πλατφόρμα, αλλά κανείς δεν υποχρεώνεται να εφαρμόζει οτιδήποτε. Σκοπός παραμένει μια ανταλλαγή απόψεων για να καταπολεμηθούν αυτές οι πρακτικές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνεργανωτή. Επειδή υπάρχει ένα, μια έντονη τάση κεντρικής διαμόρφωσης όλων αυτών των συναιτημάτων θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με διάφορες από τις προτάσεις και θα πρέπει να δούμε πώς θα δημορφωθεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Μαρίνιο Επίντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη της της εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί μια προσπάθεια την οποία θα διεξεγάγουν όλοι και η, και η Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και υπονομεύει και, την, και τα κοινωνικά συστήματα. Έτσι προκαλείται και στρέβλωση της αγοράς εργασίας και της οικονομίας της αγοράς. Ενώ δεν μπορούμε να αγγίθουμε έτσι και τα κοινωνικά ε, επιδόματα των εργαζομένων. Και πολλοί εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι, όπως οι γυναίκες, οι μετανάστες. Συχνά υπάρχουν περιπτώσεις εκμετάλλευσης των ε, ατόμων που κάνουν πρακτική. Με την πρόφαση της επαγγελματικής ε, κατάρτισης ουσιαστικά οι νέοι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και δουλεύουν με χαμηλούς μισθούς και χωρίς μισθούς. Ευχαριστώ, κύριε Λεϊερικ ανάπτυξη της αργασίας εργασίας δείχνει και καταδεικνύει την δυσλειτουργία των οικονομιών μας, των κοινωνιών μας και της γενικότερης κρίσης. Ε, όλο αυτό δείχνει πώς η λιτότητα μας προωθεί στη μαύρη εργασία. Είναι κάτι άδικο και αδικαιολόγητο για τους εργαζόμενους ε, να εργάζονται χωρίς καμία κοινωνική εξασφάλιση ε, και τραβάει προς τα κάτω ο, γενικά τις συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελεί μία έλλειψη, δημιουργεί έλλειψη σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και ε, τα έσοδα του κράτους. Και η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων επιτρέπει ακριβώς ε, την διόνυση αυτών των ε, πρακτικών. Με το νέο μοντέλο της αυταπασχα... Αυταπασχα... αυταπασχόλησης τηρούμε και πάλι τα ίδια πρότυπα. Με τα νέα αυτά πρότυπα λοιπόν δεν υπάρχει καμία κοινωνική υποχρέωση. Η πλατφόρμα που αποφασίζεται είναι μια καλή απόφαση. Όμως πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ε, αναθεώρηση της οδηγίας ε, περί απόσπασης εργαζομένων, ε, των διασυνοριακών εργαζομένων ευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασίας και ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα διαμορφώσει την προστασία, την κοινωνική προστασία και την προστασία της ασφάλειας και της απασχόλησης για όλους. Λόπε για λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Για να υπάρξει ανάπτυξη και για να είναι χρήσιμη για όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης καλύτερης ποιότητας. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία και τις συνέπειες που έχει για την κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο φύγει τους εργαζομένους, τις συνθήκες εργασίας τους, τις μισθολογικές τους συνθήκες και την συνταξιοδοτική τους διαδικασία δημιουργεί προβλήματα στα κοινωνικά συστήματα, δημιουργεί στρεβλό ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις και έτσι ε, μεγενθύνεται η υπόγεια αυτή η οικονομία. Τον τελευταίο καιρό ήρθε στην επιφάνεια πως στην Ισπανία που έχει τόσο υψηλή ανεργία λέγεται ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι αδήλωτοι, δηλαδή ένα τεράστιο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού. και δυστυχώς αυτό συνιστά ουσιαστικά εξαπάτηση και μη σεβασμό των, εργατικών, των εργασιακών ρυθμίσεων. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία και να μετατραπεί σε επίσημη απασχόληση, νόμιμη απασχόληση και μέσω των, της συνεννόησης και μέσω του ελέγχου η πλατφόρμα θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα την πραγματικότητα την οποία έχουμε να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πυρίνσκι, για την ιδιαίτερη επαγγελματική του προσέγγιση σε ό,τι φορά και τις διαπραγματεύσεις. Όμως με προβληματίζει όχι μόνο το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας, αλλά και η ανοχή της κοινωνίας ως προς αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό θα ήθελα να παροτρύνω τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν περισσότερο με την πρόληψη, αλλά και την ε, ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του, ώστε να μην γίνεται δεκτή η αδήλωτη εργασία. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και την κοινωνία σε ό,τι αφορά τι ε, επιπτώσει τη αδήλωτη εργασία. Γιατί ε, έτσι οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία κοινωνική εξασφάλιση, χαμηλούς μισθούς, στη συνέχεια χαμηλές συντάξει και από την άλλη τα κράτη-μέλη στερούνται πολύ σημαντικά έσοδα και έτσι επηρεάζεται αρνητικά και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και εν γέννη η οικονομία. Όμως τρευλώνεται και ο ανταγωνισμός. Κατά τρίτον, η αδήλωτη εργασία είναι ιδιαίτερως διαδεδομένη σε κλάδους όπου ασχολούνται ιδιαίτερως οι γυναίκες, όπως είναι η φροντίδα των ηλικιωμένων, ε, τα, ο καθαρισμός των οικοκυριών και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει έλεγχος και νομιμοποίηση αυτών των κλάδων. Όμως η εργαζόμενοι και εργαζόμενε σε αυτού του κλάδου συνήθω δεν έχουν καμία ε, δικλίδα ασφαλεία. Γι' αυτό ελπίζω η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αδήλωτη Εργασία να αποβεί αποτελεσματική και να ενισχύσει τη συνεργασία με χρήση των μελών. Επίτροπε Τάισεν, είπατε ότι θα κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να είναι αποτελεσματική αυτή η πλατφόρμα και να λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρασνοτζεύσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα που αναφέρεται στην έκθεση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου της εργασίας μόνο εάν ε, βοηθήσει και συμβάλλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μόνο εάν δεν αποτελέσει μέσω επιβολής μίας και μόνο λύσης για όλους. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τους υπερβολικούς φορολογικούς συντελεστές ε, και άλλο κόστος, άλλες, άλλα τέλη. Πρέπει να εξετάσουμε πώς αυτό συνδέεται με τις νόμιμες θέσεις εργασίας και τους ε, υψηλούς μισθούς. Ταυτόχρονα πρέπει να εξετάσουμε και το άκαμ το εργασιακό δίκαιο αλλά και τα ασφαλιστικά συστήματα και τα εξαιρετικά συστήματα που συχνά έρχονται σε αντίθεση και με τα δημοσιονομικά προβλήματα. Πρέπει να εξετάσουμε και το ζήτημα της αποδοχής ε, ε, της αντίλωτης εργασίας και μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατομελών. Ευχαριστώ κυρία Άγιος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας. Είναι κάτι το ζωτικό όχι μόνο για τα δημόσια έσοδα, αλλά και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους εργαζόμενους. Αυτά τα οποία σημαίνουν μέχρι τώρα δυστυχώς δημιουργούν προβλήματα στα δικαιώματα των εργαζομένων, στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, στα δικαιώματά τους σε συνθήκες εργασίας, στην άδεια, στην γονική άδεια και τα λοιπά, την άδεια μητρότητας, στις υπερορίες. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι είναι απελπισμένοι και αναγκάζονται να εργάζονται χωρίς να το δηλώνουν και δυστυχώς η υψηλή ανεργία ε, χτυπά ιδιαίτερα πολλές χώρες οι οποίες υποκύπτουν. Συνεπώς λοιπόν η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης και ελέγχου είναι απαραίτητη. Κυρία Κοσλόφσκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αδήλωτη εργασία είναι κάτι το οποίο κοστίζει σε επίπεδο κοινωνικό καταστρέφει την αγορά εργασίας και αρνείται να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος έλεγχος και επιθεώρηση των συνθήκων εργασίας και των συνθήκων αμοιβή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η καταπολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης είναι κάτι το οποίο περνάει και από τη μείωση των γραφειοκρατικών και οικονομικών βαρών για τους εργοδότες. Απαιτείται όχι περισσότερη νομοθετική ρύθμιση, αλλά καλύτερη νομοθετική ρύθμιση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει κυρίως για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ξέρουμε τι γίνεται με τα μπλοκάκια, με τα βάουτσερ σε χώρες όπως ε, το Βέλγιο και η δική μου χώρα και δυστυχώς απαιτείται ε, να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Απαιτείται να προετοιμάσουμε λοιπόν νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και να υπάρξουν καλύτεροι έλεγχοι και επιθεωρήσεις. Μπενιφέη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο. Θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός οργανισμού υψηλού επίπεδου με στόχο την αντιμετώπιση της υπόγειας ή μαύρης απασχόλησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα δημοσιονομικά της κάθε χώρας μέσω της μείωσης της φορολογίας αλλά κυρίως δημιουργεί προβλήματα στους εργαζομένους, στην κοινωνία, στην υγεία, στην κοινωνία γενικότερα λοιπόν, ιδιαίτερα σε τομείς όπως ο, ο, ο γεωργικός τομέας. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε τεράστιες περιοχές, ιδιαίτερα στις εύθραυτες κοινωνικές ομάδες όπως και οι μετανάστες, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι μετανάστες. Η κοινωνία των πολιτών λοιπόν μπορεί να βοηθήσει, τα συνδικάτα μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να συλλάβουμε το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος. Θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια αποκατάστασης των θέσεων αυτών απασχόλησης. Νομίζω ότι η προσπάθεια που έγινε για τη βελτίωση του κειμένου ήταν μια καλή προσπάθεια και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό τον εισηγητή Πυρίνσκι. Κυρία Τάισεν, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι οι προτάσεις τις οποίες κάνουμε να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Στίβενς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε, συνάδελφοι. Νομίζω ότι με την έκθεση αυτή κάναμε μια καλή αρχή. Και αυτό το τονίζω. Η μαύρη εργασία αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και ζημιώνει σημαντικά την οικονομία γιατί ουσιαστικά στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Και όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού για να καταπολεμήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τη μαύρη εργασία. Και ως εκ τούτου είναι καλή ιδέα να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα προκειμένου να είναι σωστή και στοχευμένη η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων. Είναι άλλωστε λογικό και απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ένα ρόλο στο συγκεκριμένο πλαίσιο και νομίζω ότι ο, ο εισηγητής τονίζει η Ένωση να σέβεται τις ε, αρμοδιότητες των κρατών μελών και να μην ξεπερνάτε τα καθήκοντά της. Ε, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει δικαίωμα να καταρτίζει νομοθεσία και να παίρνει μέτρα για τα συγκεκριμένα προβλήματα που παίρνει. Και επειδή το σέβεται αυτό λοιπόν η έκθεση, την υποστηρίζω και εγώ χωρίς ε, αμφιβολία. Ευχαριστώ, Μπιλμπάου Μπαραντίτσα, για ένα λεπτό, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να υπάρξει νομιμοποίηση των θέσεων αυτών απασχόληση των μη αναγνωρισμένων. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης, γιατί οι εργαζόμενοι είναι προσωρινοί, δεν έχουν καμία προστασία και χάνουν την αξιοπρέπειά τους. η ισχυρή αυτή ε, μαύρη θα έλεγα απασχόληση δείχνει και το μέγεθος της μαύρης οικονομίας γενικότερα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα και σε περιφερειακό προβλήμα, ε, επίπεδο. Φύγονται ιδιαίτερα οι γυναίκες, συνεπώς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και καταδικάζουν τις γυναίκες το να αντιμετωπίζονται με έλλειψη ισότητας και δικαιοσύνης. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πειρατική δραστηριότητα που υπονομεύει τα κοινωνικά μας μοντέλα. 1,5 λεπτό κυρία Ριμπέρο. Η αδίλεπτη εργασία αποτελεί ένα κοινωνικό και οικονομικό θέμα με πολύ σοβαρές συνέπειες. Υπονομεύει τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των πολιτών και έχει επίσης σημαντικές συνέπειες ε, στους προπολογισμού. Μειώνει τα φορολογικά έσοδα και επηρεάζει τα κοινωνικά δικαιώματα. Η απόφαση λοιπόν ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια πλατφόρμα για την αντιμετώπιση τη αδρέτης εργασία αποτελεί μια σωστή ιδέα και είναι απαραίτητο να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά πέρα από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών για το πώς θα προληφθούν και θα τιμωρηθούν αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να προωθηθεί και η δεδηλωμένη εργασία, η νόμιμη εργασία. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων γιατί πολλοί εργαζόμενοι εξουθούνται στην αντίλατη εργασία λόγω έλλειψης καταχώρησης και θα πρέπει λοιπόν να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις όπου ο κόσμος ε, δεν θα δουλεύει στην αντρέτη εργασία, προωθώντας την νόμιμη απασχόληση, προκειμένου και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι πολλά μπορούν να κερδίσουν από την δηλωμένη εργασία. Και θα ήθελα να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάγκη να προωθήσει τον φόρο επί των εισοδημάτων και την ε, την αρρύθμιση αυτού με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την επιβίωση στα νοικοκυριά και στις οικογένειες. τα κρατημέλη ενδεχομένως να αλλάξουν τους συντελεστές φορολόγησης γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει κίνητρο να διαφεύγει τις φορολόγησης κανείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ρέγνερ για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι οι επιχειρήσεις με γραμματοκιβώτια να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της άδελφης εργασίας. Και γι' αυτό γιατί, γιατί οι εργαζόμενοι σε περίπτωση ε, νομικής διανέξης ε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και φυσικά ανοίγει και η πόρτα για την φοροδιαφυγή. Η μαύρη εργασία είναι σκάνδαλο. Όχι μόνο οι παραδοσιακέ μορφές μαύρης εργασίας, αλλά και οι νέες μορφές ε, πλασματικής αυτοαπασχόλησης. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά μια μορφή αποφυγής των κοινωνικών προτύπων, των οικονομικών και φορολογικών προτύπων. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να εμπίπτει στο πλαίσιο της αντιλέτης εργασίας. Η πλατφόρμα λοιπόν αυτή για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας είναι σημαντική θεωρώ για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη προκειμένου να ξέρουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στην κάθε χώρα. Γι' αυτό λοιπόν ε, με αδαιμονία αναμένω τις πρώτες εκθέσεις της πλατφόρμας για να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε και τις ελεγκτικές αρχές. Και στο τέλος του δρόμου αυτού, ο οποίος ήταν μακρύς, θα ήθελα να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασίας. Thank you. Αν δεν είναι εδώ. Κύριος Γολά. Για ένα μισή λεπτό. Η αδήλωτη εργασία είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Κρίσιμο εξαιτίας της θέσης του στην παραοικονομία. Και η καταπολέμηση αυτής της αδήλωτης εργασίας είναι απαραίτητη για τα κράτη-μέλη και είναι απαραίτητο να υπάρξουν συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να γίνει αυτό. Με ενθουσιασμό και ζέση λοιπόν θα υπερψηφίσω τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. Οι αρνητικές επιπτώσεις της αδίλωτης εργασίας είναι πολυάριθμες και πολύ σημαντικές για τον προπολογισμό, τον κρατικό, για την ισορροπία του ασφαλιστικού και συστήματος και κοινωνικής ασφάλισης, για τον ε, αθέμητο ανταγωνισμό και τις επιχειρήσεις, για τους ε, εργαζομένους που χάνουν τη σύνταξή τους, την κοινωνική τους ε, περίθαλψη, και την πρόσβασή του σε μια αξιοπρεπή θέση εργασία, αλλά και στο φορά τα εργασιακά ατυχήματα. Τι σημαίνει λοιπόν ένα εργασιακό ατύχημα για έναν εργαζόμενο, η οικονομική καταστροφή και για τον εργαζόμενο που δεν είναι ασφαλισμένο, αλλά και για μια επιχείρηση, ιδίω μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε αυτή την πλατφόρμα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις επιχειρήσεις της ταχυδρομικής θερίδας και τους ε, ψευδός αυταπασχολούμενους. Δεν θα τα λύσει όλα η πλατφόρμα, όμω πρέπει να την υλοποιήσουμε, να την εφαρμόσουμε και να προχωρήσουμε με μια ευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασία για να γίνεται και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Ο ευρωπαϊκό χώρο, είμαι πεπισμένο ότι θα πρέπει να είναι ένα χώρο καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και ένα χώρο ε, κοινωνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λόπεθ, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα για την καταπολέμηση της μάστιγας της αδήλωτης εργασίας. Μια πλατφόρμα που θα επιτρέψει την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών που θα μπορέσει ίσως να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το διαρκές πρόβλημα για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στην Ισπανία αλλά και σε άλλες χώρες. Οι εργαζόμενοι είναι τα πρώτα θύματα αυτού του φαινομένου, δεν έχουν ασφάλεια στην απασχόληση, δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν κοινωνικές παροχές. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για την οικονομία μας, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για τα δημοσιονομικά μας. Είναι λοιπόν κάποια θετικά μέτρα αυτά που προτείνονται ιδιαίτερα και το θέμα των συλλογικών συμβάσεων που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, όλες οι χώρες να συμμετέχουν στην πλατφόρμα και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν ένα κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη μορφή συνεργασίας. Είναι ένα βήμα λοιπόν, πολλά όμως μένει να γίνουν, θέλουμε να ληφθούν μέτρα πιο αποφασιστικά στο μέλλον γιατί όπως είπα το πρόβλημα είναι τεράστιο, είναι μια μάστιγα για την οικονομία και την κοινωνία. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Σάντερ, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σήμερα η υπόγεια οικονομία ανέρχονται σε πολλά δις ε, κάθε χρόνο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα λοιπόν σε ό,τι αφορά την υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων, φτωχοποίηση και στέρηση σημαντικών εσόδων από τα κρατικά ταμεία και το καθεξής. Ε, αλλά και για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και 90% των επιχειρήσεων που είναι τα πρώτα θύματα. Η πλατφόρμα που υιοθετούμε σήμερα θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδίλωσης εργασίας, γιατί επιτέλους φέρνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσει σε όλα τα Θα επιτρέψει έναν σε βάθος διάλογο μεταξύ των ε, επιμέρους διοικήσεων και κυβερνήσεων και θα επιτρέψει να περιορίσουμε την ε, προσφυγή ε, στην ψευδή αυταπασχόληση και στις επιχειρήσεις της ταχυδρομικής στηρίδας. Αυτή η συνεργασία θα περιορίσει ακόμα και το δικαστικό φόρτο αυτή τη στιγμή. Όμως θα πρέπει να μείνουμε μόνο στο πνεύμα της πρότασης για αυτή την πλατφόρμα. Πρέπει να περάσουμε στην πρακτική εφαρμογή της για να επιτρέψουμε και, τις, ε, και τους ελέγχους και τις κυρώσεις. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην απάτη που συνδέεται με την απόσπαση εργαζομένων. Όμως, προσοχή, από μόνη της πλατφόρμα δεν θα κάνει τα πάντα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν και να ασχοληθούν με μια πραγματική καταπολέμηση ε, της ε, ανομίας ε, και της αποφυγής της φορολόγησης για να επιστρέψουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι στην νομιμότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάιμον για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι κάπως περίεργο το ότι η σημερινή συζήτηση για το θέμα αυτό συμβαίνει μετά τις ε, διαπραγματεύσεις, οι οποίες ήταν ε, χρονοβόρες και που ολοκληρώθηκαν μετά τον τριμερή διάλογο. Η συζήτηση λοιπόν γίνεται μετά τη διαπραγμάτευση. Αυτό μήπως ε, δεν είναι αντίρρητη εργασία από πλευρά του Κοινοβουλίου. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να απαντήσω στους συναδέλφους από το UKIP. Παρά το γεγονός ότι ο συνήθω δεν είναι εδώ για τη συζήτηση, όχι αυτή που μίλησα. Ούτε αυτοί που μίλησαν δεν κάθισαν να ακούσουν την υπόλοιπη συζήτηση. Έκαναν το θέατρο τους και μετά σηκώθηκαν και έφυγαν, ως συνήθως. Πολλές ανώσεις ακούσαμε για το ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μέτρα γιατί είναι κατά του ανταγωνισμού. Προσπάθησαν να μας κάνουν και μάθημα για την ανταγωνιστικότητα και ως συνήθως δεν καταλαβαίνουν ούτε τα οικονομικά ούτε τον ανταγωνισμό. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το άκρο της αγοράς εργασίας χρειάζεται ρύθμιση προκειμένου να υπάρχουν ίσοι όροι και αυτοί που υποφέρουν από την νομοθεσία αυτή είναι ακριβώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίοι δεν έχουν ανταγωνισμό από τις μεγάλες πολυεθνικές, αλλά από τους μικρούς που δεν πληρώνουν φόρους και έτσι έχουν παράνομα πλέον εκτήματα. Και αν καταλαβαίνετε τίποτα θα καταλαβαίνετε και αυτό. Κύριε Σούλτσα για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σήμερα πολλά παραδείγματα ακούσαμε για την καταπολέμηση της ε, άντρα τη εργασίας και γιατί είναι τόσο σημαντική και για τα κράτη-μέλη αλλά και για τους ε, πολλούς ε, εργαζομένου. εργαζομένους. Και ένα θέμα λοιπόν είναι αυτές οι επιχειρήσεις ταχυδρομικής θηρίδα και κοιτώντα τα αριθμητικά στοιχεία για την αδηλέτη εργασία 24,6 ε, στην Ελλάδα του ΑΕΠ αλλά και στην Ιταλία και στην Γερμανία πολλά θα πρέπει να γίνουν. Είμαστε στο 13% σε σχέση με το ΑΕΠ η αντρική εργασία. Έχουμε πολλά θετικά παραδείγματα. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, λιγότερο από 10% και η δημιουργία μιας πλατφόρμας με δεσμευτική ανταλλαγή απόψεων αποτελεί κατά τη γνώμη μου ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα και μιλάμε για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να να εντοπίσει αυτή και η Επιτροπή, αυτή η πλατφόρμα, τις βέλτιστες πρακτικές και να τις υποστηρίξει για να υπάρξει εναρμόνιση και των μεθόδων καταπολέμησης και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε σύγκληση. Και σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή απόψεων, η ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών και όχι ο δεσμευτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι είναι σωστή η λύση που βρέθηκε με το Συμβούλιο και θα συνεχίσω να την υποστηρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Σόγκορ για ένα μισή λεπτό. Σα ευχαριστώ. Παρά τον ανταγωνισμό που προκαλεί και την, τον οικονομικό αντίκτυπο, η ατλέτη εργασία δεν έχει λάβει ακόμα την, προστασία, την ε, προσοχή που θα έπρεπε να έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποια προφανή εξήγηση για την δυναμική της αδρέτης εργασίας. Για παράδειγμα, αντίθετα με αυτό που θα περίμενε ο κόσμος, η αδρέτη εργασία δεν αυξάνεται σε περίοδους λιτότητας και δεν ε, επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση της φορολογίας, για παράδειγμα. Ωστόσο, αυτό που είναι σαφές από τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι ότι υπάρχουν κάποια κρατημέλη που είναι πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Η αντίληπτη εργασία για την Αυστρία, για παράδειγμα, είναι, για παράδειγμα, πέντε φορές πιο κάτω από ό,τι στη χώρα μου. Αν με την πλατφόρμα αυτή λοιπόν καταφέρουμε να μεταφέρουμε μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ τομέων κάποιες από τις βέλτιστες πρακτικές και να ρυθμίσουμε έτσι την αγορά, αυτό όχι μόνο θα προωθήσει τον θεμητό ανταγωνισμό και την, ε, τα δημοσιονομικά, αλλά θα βάλουμε και τέλος την εκμετάλλευση εκατομμυρίων εργαζομένων που δεν έχουν ε, επιδόματα και συνταξιδιτικά δικαιώματα. Επίσης, θα καταφέρουμε να ε, δώσουμε μεγαλύτερο ένασμα και στην εμπιστοσύνη του κόσμου στην ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Φαντεκάντελάρε για 1,5 λεπτό. Επιτροπέ, συνάδελφοι, η αθέμητος ανταγωνισμό στην αγορά εργασία υπονομεύει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο ευρωπαϊκό project. Και με την ίδρυση λοιπόν τη πλατφόρμα, η Ευρώπη κάνει ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση τη αντίλωτη εργασία, τη πλασματική αυτοπασχόληση και ούτω καθεξής. Και θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού, αλλά η απάτη ασφαλώ δεν σταματάει στα εθνικά σύνορα και γι' αυτό είναι καλό που αναλαμβάνει τι ευθύνε τη και η Ευρώπη. Η ευθύνη που έχουμε για τους εργαζόμενους ε, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Και αυτό κυρίως ε, επηρεάζει τις ευάλωτες ομάδες όπως οι γυναίκες, όπως οι μετανάστες, αλλά και ευθύνει έναντι των κρατών μελών, τα οποία χάνουν έσοδα με τις απάτες αυτές. Η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπονομεύεται. Γι' αυτό λοιπόν η λέξη κλειδί είναι συνεργασία και γι' αυτό λοιπόν ζητώ να μην ε, οξυνθούν οι διαφορές μεταξύ των χωρών της ε, Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν και στις επιθεωρήσεις εργασίας και θα ήθελα να τονίσω πόσο αναγκαίο είναι να υπάρξει περαιτέρω ψηφιοποίηση των δεδομένων όπως το εσωτερικό το σύστημα εσωτερικής αγοράς και πληροφόρησης. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν αποτελεί σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και πολύ παραπέρα. Και γι' αυτό λοιπόν με αδειμονία περιμένω και το πακέτο για την κινητικότητα της εργασίας από την Επιτροπό Τέισεν. Ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε στην διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Ο κύριος Χάτμαν, πρώτος ομιλητής. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η αδήλωτη εργασία και η πλασματική απασχόληση επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη. Και παρότι τα περισσότερα στοιχεία αφορούν ε, την πρόληψη και αποτροπή, είμαι πεπισμένος ότι και οι ευρωπαϊκές ε, ενέργειες θα είναι ε, ευπρόσδεκτες και αποτελεσματικέ πέραν του εθνικού πλαισίου δηλαδή. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και επηρεάζει μάλλον αρνητικά τον επαγγελματικό και προσωπικό βίο πολλών Ευρωπαίων. Η συνολική φύση αυτού του φαινομένου και η διευρυμένη του παρατήρηση δείχνει ότι μόνο από κοινού μπορούμε ε, να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο και όταν καταπολεμούμε όλες τις πτυχές του. Πάντα βεβαίως ε, σεβόμενοι και την ε, αρχή της επικουρικότητας. Επίσης, θεωρώ θετικό ότι συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι ως ισότιμα μέλη. Ελπίζω λοιπόν αυτή η πλατφόρμα να αποτελέσει χώρο ισότιμης συνεργασίας και κατάρτισης ολοκληρωμένων στρατηγικών. Ευχαριστώ κυρία Αρπίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Επίτροπε, η έκθεση αυτή είναι μια, ένα θετικό βήμα. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά είναι καλό που το κάναμε. Ευχαριστώ λοιπόν και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές δεν θα ήθελα τώρα να υπενθυμίσω και εγώ με τη σειρά μου τις αρνητικές συνέπειες της παράνομης εργασίας και φυσικά δεν θα ήθελα και εγώ να υπενθυμίσω τις αρνητικές συνέπειες για τα δημοσιονομικά των κρατών μελών. Είναι απαραίτητο λοιπόν τα μέτρα τα οποία προτείνονται να ελεγχθούν σύντομα, να δούμε τι αποδίδουν και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό γρήγορα η, η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών είναι κάτι το χρήσιμο. Νομίζω όμως ότι η μορφή αυτής συνεργασίας την οποία προτείνουμε που είναι θετική δεν είναι από μόνη της ικανή να αναστρέψει το φαινόμενο αυτό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την συνειδητοποίηση των εργοδοτών και των εργαζομένων έτσι ώστε να απορριφθεί πλέον το φαινόμενο. Κυρία Σαΐτοδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ενιαία αγορά απαιτεί για να λειτουργήσει κάποιους ελάχιστους κανόνες οι οποίοι να σέβονται τις βασικές μας αρχές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά στις χώρες μέλη αλλά αφορά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μου, η Τσεχία, υποφέρει από το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο. Ε, νομίζω ότι η αδήλωτη εργασία αντιπροσωπεύει πάνω από το 18% και νομίζω ότι η κοινή αυτή πλατφόρμα θα στηριχθεί και από την τσεχική κυβέρνηση, δεν επιβαρύνει με περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να γνωρίζουν το τι συμβαίνει γύρω τους για να καταπολεμήσουν αυτές τις αρνητικές τάσεις. Μείωση του κόστους της πλατφόρμας αυτής είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ο κ. Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αδήλωτη εργασία είναι συνηφασμένη με όλη τη διαδικασία απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων είναι συνηφασμένη με την τεράστια ανεργία η οποία υπάρχει και την πίεση εκ μέρους των εργοδοτών να υπάρχει μαύρη εργασία. ταυτόχρονα αδήλωτη εργασία σημαίνει και τεράστια απώλεια εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό το βλέπουμε ειδικότερα στην ελλάδα που έχουμε μια τεράστια εισφοροδιαφυγή μια εισφοροδιαφυγή η οποία υπονομεύει την όλη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος. κατά την άποψή μου βεβαίως εάν θέλει το κράτος μπορεί να χτυπήσει την εισφοροδιαφυγή διαφυγή και αυτό μπορεί να το κάνει αποτελεσματικά. επομένως θεωρώ βέβαια σημαντική την αναγνώριση του προβλήματος σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης θεωρώ σημαντικό το ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα και η ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά είναι μια αρμοδιότητα καθαρά του εθνικού κράτους και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για να υπάρξει πραγματικά χτύπημα της αδήλωτης εργασίας και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λυκιώτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αδήλωτη εργασία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για ολόκληρη την Ένωση. Δεν πρέπει όμω σε καμία περίπτωση να μπερδεύουμε την αδήλωτη εργασία με τη φοροδιαφυγή. Τα μνημόνια, οι πολιτικέ λιτότητα, τα ψηλά ποσοστά ανεργία επιβαρύνουν τους πολίτες και σπρώχνουν πολλούς εργαζόμενους στην επισφάλεια με τις επιχειρήσεις να στηρίζουν αυτή την πρακτική και να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους εργαζόμενους και πολλά κράτη μέλη να κλείνουν τα μάτια. η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασία μπορεί να είναι βοηθητική χωρίς να αντικαθιστά τις εθνικές αρχές εργασίας και εμάς μας βρίσκει σύμφωνους ως αριστερά όμως η λύση για την καταπολέμηση της αδείλωτης εργασίας αλλά και του ντάμπινγκ μισθών πρέπει να λυθεί μόνο όταν τα κράτη μέλη ορίσουν προστατευτικούς νόμους υπέρ των εργαζομένων όταν κατοχυρώσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. επίσης για μας πρέπει να ανατραπούμε τις κινητοποίησεις των εργαζομένων οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκληρής λιτότητας και τα μνημόνια τα οποία σπρώχνουν τους εργαζόμενους στη φτώχεια και στην επισφάλεια της εργασίας τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστούμε. Έχουν ζητήσει και άλλο το λόγο, αλλά θα σταματήσουμε εδώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επιτροπέ Ναι, κύριε Θρέτς. Συγγνώμη, διορθώστε με αν σφάλω. Αλλά νόμιζα ότι η διαδικασία προβλέπει ότι όταν υπάρχουν πολλοί στο Catch the Eye θα έχουμε έναν από κάθε ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει πάρει το λόγο μου κάποιος από το EFTD. Κύριε Εύριτζ, από ό,τι ξέρω αναπόκειται στον πρόεδρο να αποφασίσει εξαρτάται και από τον χρόνο ε, της ίδιας της συζήτησης. Σήμερα ε, δώσαμε το λόγο σε όσους ήθελαν να πάρουν το λόγο με την μπλε κάρτα και έτσι αυτό μας επηρεάζει και στο χρονικό μας περιθώριο. Ε, δεν είναι απαραίτητο να δώσω το λόγο σε κάθε πολιτική ομάδα. Προσπάθησα να είμαι δίκαιη γιατί σε εσά, α πούμε, δεν πήρατε το λόγο τώρα, αλλά πήρατε πριν μπλε κάρτα. Επομένω, νομίζω ότι συμμετείχατε και σε επαρκώ στη συζήτηση. Επίτροπε Τέσσερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Σήμερα θα εγκρίνεται την απόφαση για την ε, αντιμετώπιση της ε, μαύρης εργασίας, της εργασίας και αύριο θα ψηφίσετε και για το πακέτο το φορολογικό, για το οποίο θα κάνετε και συζήτηση μάλιστα. Και οι δύο φάκελοι ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Ε, πρόκειται για πρωτοβουλίε που θα καταστήσουν σαφέ ότι η Ευρώπη είναι μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινέ αξίε και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Και οι δύο φάκελοι θα μεριμνήσουν και η πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία ότι θα υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τον επιχειρηματικό βίο και ιδίω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι ο καθένας συμβάλλει σε δίκαιο βαθμό και στη φορολογική πολιτική και ότι η αδήλωτη εργασία θα καταπολεμάται και κατά προτίμηση θα μετατρέπεται σε νόμιμε και αξιοπρεπεί θέσει απασχόληση, κάτι το οποίο είναι καλύτερο για όλου. Αξιότιμα μέλη. Η πλατφόρμα αφορά όλε τι ενδιαφερόμενε αρχέ και του κοινωνικού εταίρου και αυτό είναι θετικό να έχουν και αυτή μια φωνή, γιατί εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τον καθένα την ε, πραγματικότητα στην πράξη. Η πλατφόρμα παρέχει μία δομή, αλλά χωρίς υποχρέωση ε, για μία διασυνοριακή προσέγγιση που είναι και πολύ αποτελεσματική. Η πλατφόρμα αντικαθιστά, δεν αντικαθιστά τις ε, επιθεωρήσεις από τα κράτη-μέλη, ούτε αφαιρεί τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Απλώς ε, διευκολύνει τη συμπλήρωση των μέσων που έχει διαθεσή του το κράτος μέλος και θα κάνει συστάσεις ε, προς τα κράτη-μέλη να γίνουν πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και να γίνει και μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί όχι. Με μια κοινή συνεργασία λοιπόν αυτό θα, θα όλοι και δεν το λέω μόνο εγώ, άκουσα ότι και εσεί το λέτε. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ούτω ώστε να στηρίξουμε στον απαραίτητο βαθμό την πλατφόρμα και βεβαίω, όπως έχει συμφωνηθεί ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο και θα υποβάλουμε εκθέσεις. Και σε ό,τι φορά το πακέτο κινητικότητας, το οποίο δεν είναι το σημερινό μας ε, ζήτημα και αντικείμενο, αλλά έχουν τεθεί διάφορα ερωτήματα, για το πακέτο κινητικότητας ε, ελπίζω, όπως και πολλοί από εσά, γρήγορα να έχουμε τις πολιτικές συγκυρίες και συνθήκες για να ξεκινήσουμε και αυτό το ζήτημα, γιατί και αυτό το πακέτο κινητικότητας ε, χρειάζεται ίσους όρους ανταγωνισμού και κοινωνική δικαιοσύνη πέραν της ε, διευκόλυνσης της εργασιακής ε, κινητικότητας που είναι απαραίτητη στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι τον εισηγητή και όλους τους διαπραγματευτές που συμμετείχαν στους τριμερείς διαλόγους και προσβλέπω σε θετικά αποτελέσματα μαζί με όλους εσά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Για να συνοψίσουμε τη συζήτηση, έχει το λόγο ο κύριος Πυρίνσκι, εισηγητής. Παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση επιτέλεσε έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Όπως ανέφερε και η κυρία Επίτροπος στην πρωτολογία της, είναι ιδιαίτερα σοβαρό και σύνθετο το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας. Και υπάρχει αντίστοιχα μεγάλη ανάγκη για ξεκάθαρη και αποτελεσματική και ρητή αναφορά σε αυτά τα προβλήματα, στον προσδιορισμό τους και στην ε, ε, διαμόρφωση κοινών λύσεων. Θα ήθελα και εγώ να επισημάνω και είναι το συμπέρασμα που απορρέει ότι οι πολλές άμεσες επιπτώσεις της αδίλωτης εργασίας στους εργαζόμενους, στα φορολογικά συστήματα, στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και στον ανταγωνισμό ουσιαστικά αποτελούν απειλή στον ίδιο τον κοινωνικό ιστό σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν κάνω λάθος, χθες το βράδυ ο πρόεδρος Δράγκη ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφέροντας ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει όλο ένα και περισσότερες παραβάσεις σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής και οικονομικής συνοχής. Και δεν είναι τυχαίο που ξεκίνησε, θεωρώ την παρέμβασή του. Γιατί όσο και αν καταβάλουμε προσπάθειες για την ε, απασχόληση, για την φορολογική πολιτική και το καθεξής, αν ο ίδιο ο κοινωνικό ιστός στον οποίο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα καταστρέφεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχουν τα υπόλοιπα μα μέτρα. Γι' αυτό κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι τα όσα έχουν αναφερθεί για αυτή την πλατφόρμα και από ό,τι καταλαβαίνω και από τις παρεμβάσεις, η πλατφόρμα λοιπόν έχει ε, επιτύχει μία ισορροπία μεταξύ των ε, συμφερόντων των κρατών μελών αλλά και της Ένωσης από την άλλη για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος. Δεν έχω άλλο χρόνο, μπορώ μόνο να συμφωνήσω με τα όσα αναφέρθηκαν ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί πριν από το καλοκαίρι και ε, στηρίζω και τις δηλώσεις της κυρίας Τάισεν, της Επιτρόπου και να ξαναφέρουμε ξανά και ξανά αυτό το ζήτημα στο Κοινοβούλιο και στην Ολομέλεια, γιατί είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη συζήτηση ε, και ε, ανάληψη δράσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι. Κλείνει η συζήτηση.